So colleagues could maybe, maybe take Συνάδελφοι παρακαλώ καθίστε για να αρχίσουμε την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης. Συνάδελφοι και φίλοι, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί σήμερα εδώ στις Βρυξέλλες έχουμε κοντά μας έναν, τον δόκτορα Ντένις Μοκουέγγε που έχει τιμηθεί με το βραβείο Σαχάροφ του 2014. Ο δόκτωρας Μακουέγγι είναι εξαιρετικός άνθρωπος που διευθύνει ένα εξαιρετικό νοσοκομείο στο Κονγκό, το επισκέφθηκα και εγώ πριν από ένα μήνα και είδα τη δουλειά που κάνει σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες φροντίζει γυναίκες και παιδιά που είναι θύματα βιοπραγιών και της σύραξης στο Ανατολικό Κονγκό, στα ανατολικά του Κονγκό. Ο Δόκτωρ Μακουέγκε προσήλθε σήμερα για να μας μιλήσει για τα προβλήματα στο ανατολικό τμήμα του Κονγκό και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν εκείνο το μέρος του κόσμου και που αφορούν και την ανάπτυξη. Η Επιτροπή μας κύριε Μακουέγγι, φροντίζει για την αναπτυξιακή βοήθεια από την Γενική Διεύθυνση ΕΦΚΟ αλλά και για την ανθρωπιστική βοήθεια και ξέρω ότι στο νοσοκομείο στο Πάντζι είχαμε μιλήσει για το ότι η Ένωση ήδη βοηθάει το νοσοκομείο και το Ίδρυμά σας και γενικά σας βοηθάει. Θέλουμε λοιπόν να σας ακούσουμε για τη δουλειά που κάνει το Ίδρυμα και το νοσοκομείο σας και γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολη η καιρή στο Ανατολικό Κονγκό και στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Προβλέπονται εκλογές στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, στο Μπουρούντι και στη Ρουάντα τους επόμενους μήνες. Στο Μπουρούντι θα ξέρετε από τις εφημερίδες ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή διότι ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θέλει να είναι υποψήφιος για τρίτη φορά και προβλέπονται και τοπικές και περιφερειακές εκλογές για μετά λίγους μήνες και μετά εθνικές το 16 και στη Ρουάντα επίσης. Είναι λοιπόν περίοδος πολιτικής αβεβαιότητας και εμείς ελπίζουμε ως ευρωβουλευτές να μπορέσουν να γίνουν οι εκλογές σε ήρεμο πνεύμα αληθινής δημοκρατίας όπου θα πριτανεύσουν και θα προωθηθούν τα συμφέροντα των πολιτών. Ξέρω, δόκτωρ Μακουέγγι, ότι το Νοέμβριο όταν μιλήσατε στο κοινοβούλιο ο λόγος σας ήταν πολύ συγκινητικός και από τότε που δεχτήκατε το βραβείο αντιμετωπίσατε γνωρίζω και προσωπικές δυσκολίες και αφισβητήθηκε και η ασφάλειά σας εκεί στο Κονγκό. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που μπορέσατε να έρθετε για να συμμετάσχετε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ε, μάλλον και στις ε, ημερίδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την κυρία Λούνατσεκ και χαίρομαι και για τη δική της παρουσία. Σήμερα έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανάπτυξης και με εκπροσώπους των ΑΚΕ της Ισομερούς Συνέλευσης δηλαδή όπως τον Λουί Μισελ που είναι πρόεδρος της και θα του ζητήσω να λάβει το λόγο πριν τον δώσω στον κύριο Μακουέγγι. Ορίστε Λουί Μισελ μου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητέ Δόκτωρ Μοκουέγγε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Ο Δόκτωρ Μοκουέγγε είναι γνωστός. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένα υπόδειγμα θάρρους που, τον οποίο σέβονται όλοι. Είναι ένας από τους μεγάλους μάρτυρες του αιώνα μας και από τα πυλώνες της ιστορίας που έλεγε και η Μαργαρίτα Γιουρσενάρ. Το έχω ξανααναφέρει, την έχω ξαναφέρει αυτή τη φράση αλλά δεν μπορούσα να την παραλείψω και τώρα. Ο δόκτωρ Μουκέγγε έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει το σκότος και το σκοταδισμό και να προωθήσει την ζωή και τους περιφρονεμένους. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει, αλλά Μόλις πήρα ένα βιβλίο που μόλις εκδόθηκε, «Οι 100 ήρωες του αιώνα». Δεν ξέρω, Διονύση, εάν το ξέρεις, αλλά είσαι και εσύ μεταξύ τους. Μεταξύ των 100 ηρώων του αιώνα. Και αυτό το βρήκα πολύ πρέπον και έχει πάρει και άλλα βραβεία και πράγμα που δείχνει τι εκπροσωπεί είναι πάστορ, χειρούργος, γυναικολόγος, ιδρυτής και διευθυντής του νοσοκομείου Πάντζη στον Μπουκαβού και ένας πραγματικός ανθρωπιστής που τιμάει την Αφρική και τον κόσμο. Έχει κυρίως την τεράστια δυνατότητα να ακούει τον λόγο των πιο αδύναμων, των πιο φτωχών των γυναικών που έχουν υποστεί σεξουαλική βία, των καταφρονημένων γενικότερα που δεν έχουν ελπίδα και μέλλον και όπως λέει και ο ίδιος καμιά φορά εκείνων που δεν έχουν καν ύπαρξη. Γιατρεύει καρδιές και σώματα και αναζωογονεί την φλόγα που υπάρχει στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Όπως είπε και ο Αϊνστάιν, η αξία ενός ανθρώπου έγκυται στη δυνατότητά του να δίνει και όχι στη δυνατότητά του να παίρνει. Ο δόκτωρ Μουγέγκε είναι από αυτούς που δίνουν και δίνονται για να θριαμβεύσει η ζωή κατά του θανάτου, το φως κατά του σκότους, κατά της βίας, κατά της αδικίας και της ατιμορρησίας. Χάρη στην κινητοποίηση που κάνει της κοινωνίας των πολιτών και των νομικών συμβουλών που χορηγεί κινητοποιεί τις συνειδήσεις σε, μια σε ένα δίκαιο αγώνα με μεγάλη πυθό που αναγκάζει την ε, διεθνή κοινότητα να μην μπορεί πια να κλείσει τα μάτια της σε αυτά που γίνονται στο Ανατολικό Κονγκό. Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι είναι και επιστήμον ιατρός δηλαδή είναι και άνθρωπος με μεγάλη θρησκευτική πίστη αλλά πάνω απ' όλα ένας μάρτυρας που τολμά να αντιμιλήσει στους πολιτικούς και οι πολιτικοί καμιά φορά τον κατηγορούν ότι πολιτικοποιεί τα πράγματα. Αυτός δεν κάνει, δεν ασκεί πολιτική. Απλώς εκφράζει το ανθρώπινο του καθήκον ως ανθρώπου που δρά ως μάρτυρης όσων γίνονται στην κοινωνία του και ενοχλεί τη συνείδηση ορισμένων αρχών και πρέπει να σου πω Διονύση ότι κατά κάποιον τρόπο ξυπνάτε και τις δικές μας συνειδήσεις. Πολύ σημαντικό και αυτό. Διότι εμείς εύκολα εκφράζουμε προφορικά τα αισθήματά μας υπέρ των αδυνάτων αλλά εσείς το κάνετε στην πράξη και μας ταράζετε και μας τη συνείδησή μας. Ξέρετε ότι με το βραβείο Σαχάροφ όλοι σας υποστήριξαν εδώ στο Κοινοβούλιο, το οποίο και εσείς αρκετά γνωρίζετε. Και θα συνεχίσουμε και εμείς τον αγώνα δίπλα σας. Νομίζω ότι πρέπει παραπάνω από ποτέ να σας ευχηθούμε να έχετε όλο και περισσότερη στήριξη για να μπορέσετε πραγματικά να αλλάξετε τη ζωή και την πραγματικότητα και την τύχη αυτών των γυναικών που έχουν πια γίνει σαν ένας μοχλός ή αντικείμενο του πολέμου και σας συγχαίρω, ας μην μακρηγορήσω κι άλλο, εξ ονόματος όλων των κοινοβουλευτικών απλώς, θα ήθελα να σας βεβαιώσω για την, τον θαυμασμό και την υποστήριξή μας καθώς και για τα αδελφικά μας αισθήματα. Σας ευχαριστώ. Ακούσατε συνάδελφοι, έχετε ξαναδεί τον Δόκτωρ Μακουέγγι, θα του δώσω τώρα το λόγο για να μας πει περισσότερα για την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και για το πώς θεωρεί ότι μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε εδώ να υποστηρίξουμε την καταπληκτική εργασία του Ιδρύματός του. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν που με υποδέχεστε σε αυτή την έκτακτη σύνοδο της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένο. Γιατί, όπως είπε και ο Λουί Μισελ, συγκινήθηκα από την αλληλεγγύη σας, από τη διάθεσή σας να σταθείτε στο πλευρό μας, σε μία μάχη όπου συχνά αισθανόμαστε μόνοι και που είναι πολύ δύσκολο να διεξάγουμε μερικές φορές. Υπάρχει εκφοβισμός, Υπάρχει μόνιμη απειλή. Εμείς απλώς κάνουμε το καθήκον μας. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τις γυναίκες που είναι θύματα σεξουαλικής βίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και το κάνουμε γιατί έχουν τη θέση τους στην κοινωνία μας, το ξέρουμε αυτό. Και γιατί αυτή η θέση την αξίζουν. Γιατί δεν υπάρχει Κονγκό χωρίς το 50% του πληθυσμού του που αποτελείται από αυτές τις νεαρές γυναίκες, νεαρές κοπέλες και γυναίκες. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη χωρίς ειρήνη ή σταθερότητα. Μπορούμε να κάνουμε πολλές προσπάθειες, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά χωρίς ειρήνη ή σταθερότητα δεν υπάρχει ανάπτυξη. Η ασφάλεια και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι προϋπόθεση εκ των αν θέλουμε να πετύχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Στη χώρα μου, το 2013, είχαμε πολλές ελπίδες όταν υπογράφτηκε η Συμφωνία Πλαίσια της Αντίσα Μπέπα για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο Επρόκειτο για μια πολιτική και διπλωματική δέσμευση τη διεθνούς κοινότητα, για να αντιμετωπιστούν οι βαθιέ αιτίε της αστάθειας που επηρεάζει τα ανατολικά του Κονγκό εδώ και πάνω από δύο δεκαετίε. Συνδυάστηκε με μια στρατηγική για την ειρήνη και την ανάπτυξη με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας Ενώ τότε λοιπόν αισθανθήκαμε μια κάποια ελπίδα, σήμερα αυτή η συμφωνία υποσκάπτεται από δύο πράγματα. Καταρχάς, μια επιδείνωση της ε, κατάστασης της ασφάλειας, όπως είπε και η Πρόεδρος μόλις τώρα, αλλά υπάρχει και ένα προεκλογικό πλαίσιο που είναι εκρηκτικό. Καταρχάς, για το θέμα της ασφάλειας. Τα ανατολικά του Κονγκό σπαράζονται από συγκρούσεις και από πολυάριθμες ε, πολιτοφυλακές, ντόπιε και ξένες, όπου σπέρνουν τον δρόμο στις τεράστιες εκτάσεις της χώρας, όπου δυστυχώς η κρατική εξουσία είναι ανύπαρκτη. Η εξουδετέρωση των ένοπλων δυνάμεων στα ανατολικά της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό με προτεραιότητα της FDL και της ADF Ναλού σε καμία περίπτωση δεν έχει επιτευχθεί εξαιτία τη έλλειψη συνεργασία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και των δυνάμεων της Μονούσκου, που είναι η αποστολή του ΟΗΕ για την σταθεροποίηση της ανατολική περιοχής του Κονγκό. Τον Ιανουάριο του 2015, οι ένοπλες δυνάμεις του Κονγκό ξεκίνησαν μια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του FDLR χωρίς την ε, στήριξη της ε, ταξιαρχίας παρέμβασης Μονούσκο, η οποία είχε εμπλακεί μήνες στον σχεδιασμό των επιχειρήσεων. Λόγω του σεβασμού της πολιτικής ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η Μονούσκο δεν μπορεί να στηρίξει τις δυνάμεις των οποίων οι αξιωματικοί κατηγορούνται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, αυτό είναι ένα πρότυπο του ΟΗΕ που πάντα τηρείται. Εμείς ως πολίτες δεν καταλάβαμε τίποτα πάντα, θα να σας το πω. Εμείς έχουμε πολλούς αρχηγούς, οπλαρχηγούς, διοικητές κτλ. Πώς είναι δυνατόν με τόσους ε, στρατιωτικούς ε, διαλέγουμε αξιωματικούς οι οποίοι έχουν βρώμικα χέρια. Ακόμη και αν υπήρχαν υποψίες, νομίζω ότι θα, υπήρχαν, ε, θα είχαμε τη δυνατότητα να λύσουμε ειρηνικά ε, το θέμα αυτό, για να μπορέσουμε να αφήσουμε την ομάδα αυτή να κάνει τη δουλειά της, την οποία περιμέναμε. Η ADF Ναλού είναι μια πολιτοφυλακή που ανήκει στην, στον τζιχαντιστικό κίνημα Al-Shabaab και σπέρνει τον δρόμο στο Βόρειο Κιβού. Την περασμένη εβδομάδα η ταξιαρχία παρέμβασης του ΟΗΕ ε, έπεσε θύμα δύο φορές στην περιοχή του Μπενί και κάποιοι κυανόκρονοι σκοτώθηκαν στα πλαίσια της εντόλης που είχαν λάβει από το Συμβούλιο Ασφαλείας να προστατεύσουν τους αμάχους. Την ε, νύχτα της ε, Παρασκευής προς Σάββατο της περασμένης εβδομάδας, 7 άτομα σκοτώθηκαν με αχέμαχο όπλο από μέλη αυτής της πολιτοφυλακής και έτσι ο αριθμός των αμάχων που σκοτώθηκαν σε, την σε αυτό το χώρο ε, φτάνει τα 300 άτομα σε λιγότερο από 5 μήνες από τους τρομοκράτες αυτούς του αντεέθναλου. Όταν εγώ πήρα το βραβείο Ζαχάροφ είχα μιλήσει για τη σφαγή αυτή που διαπράττουν σε αυτή την περιοχή οι πολιτοφύλακες αυτοί. Και δυστυχώς από τότε έρχομαι ξανά εδώ μπροστά σα με αντίστοιχε πληροφορίε. Μα επηρεάζει πάρα πολύ το γεγονό ότι αυτή η ομάδα εν πάση αντιπορησία, συνεχίζει να σκοτώνει. Ό,τι μπορέσαμε να κάνουμε για να τι ε, παρεμποδίσουμε ε, απέδει άκαρπο. Είναι επιτακτικό από τη μία Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τι προσπάθειε στήριξη στι αρχέ τη λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για να υπάρξει μια βαθιά μεταρρύθμιση του τομέα τη ασφάλεια, που θα συμπεριλαμβάνει το στρατό, την αστυνομία, τη δικαιοσύνη και το σοφρονιστικό σύστημα και από την άλλη οι ένοπλες δυνάμεις και η Μονούσκο θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να θέσουν τέλος σε αυτές τις σοβαρότητες παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου και να σπάσουν τον κύκλο της βίας. Πάρα πολλά μέσα χρησιμοποιήθηκαν, πάρα πολλές προσπάθειες καταβλήθηκαν, αλλά δυστυχώς όταν έχουμε ένα στρατό και μια αστυνομία που δεν δρούν για να προστατεύσουν τους αμάχους, δεν υπάρχει λύση. Πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση και να υπάρξει βαθιά μάλιστα μεταρρύθμιση του στρατού και της αστυνομίας. Θεωρούμε ότι είναι ένα από τα κλειδιά για να επιτρέψουμε να επανέλθει η ασφάλεια στην περιοχή αυτή και να αρχίσουμε να μιλάμε για την ανάπτυξη. Σε εκλογικό επίπεδο το Κονγκό και οι γειτονικέ χώρε μπήκαν σε μια προεκλογική περίοδο που θα κρατήσει τρία χρόνια. Οι κατολογίε γύρω από την σταθεροποίηση των καθεστώτων που ισχύουν αυτή τη στιγμή ε, υποσκάπτουν τη δημόσια συζήτηση και δημιουργούν άγχο στου ε, πολίτε. Οι πολίτε θέτουν πολλά ερωτήματα. Μερικέ φορέ υπάρχει σιωπή και πιο πρόσφατα Κάποιοι πρόεδροι παρουσιάζονται σε εκλογές, ε, αλλά δρούν ενάντια στο Σύνταγμα. Η θέληση των ε, ηθινόντων επί, τους ε, καθυλώνει στην εξουσία ε, και υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί νέος κύκλος αστάθειας. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό το προεκλογικό χρονοδιάγραμμα αμφισβητείται από διάφορους και μία βιαστική αποκέντρωση, ενώ είχαμε πάρα πολύ χρόνο να την κάνουμε, 10 χρόνια. Τώρα ξαφνικά όμως πρέπει να την κάνουμε μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια. Και έχουμε και μία σειρά από εκλογικές αναμετρήσεις ε, να οργανώσουμε ταυτόχρονα. Όλο αυτό δημιουργεί ένα κλίμα έτσι ε, υποψίας ότι θα έχουμε καθυστερήσει στις εκλογές. Ε, φυσικά μας ανταπαντούν ότι δεν ήταν δυνατό να γίνουν ταυτόχρονα όλα και ότι δεν γίνεται αλλιώ, πρέπει να υπάρξουν καθυστερήσει κτλ καθώς πλησιάζουν αυτές οι εκλογές, το γενικό κλίμα αυτή σε αυτή την περιοχή ε, από εντάσεις, από πολιτική βία και από παραβίαση της ελευθερίας. Από την Κινσάσα μέσα στην Μπουζουμπούρα η καταπίεση των, ε, των διαδηλωτών που ζητούν την ε, αλλαγή και τη δημοκρατική εναλλαγή ε, έχει πολύ σοβαρότατα προβλήματα, παρουσιάζει πολύ σοβαρά τα προβλήματα. Κάθε μέρα έχουμε νεκρούς. Μην ξεχνάμε τι έγινε το 1993 στη Ρουάντα. Ε, προσπαθούμε ακόμα να διαχειριστούμε τις συνέπειες εκείνης της κατάστασης ε, στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Οι απειλές που υφιστάμεθα, οι εκφοβισμοί, αλλά και οι συλλήψεις πολλών ακτιβιστών στην ΣΑΣΑ, στην κόμμα, οι οποίοι κρατούνται ακόμα πολλοί από αυτούς. Μόνο και μόνο γιατί ζητούν ειρηνικά να υπάρξει μια δημοκρατική αναλλαγή στην εξουσία της χώρας τους. Πρόσφατα η κυρία Φατού Σάουντα, που είναι εισαγγελέα ε, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, μίλησε για την ανησυχία της, για αυτή την κλιμάκωση βίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία έρευνα των των εγκλημάτων που αφορούν την αρμοδιότητα του δικαστηρίου. Κυρίες και κύριοι, μηνύματα αγερμού χτυπάνε κόκκινο, αλλά δεν υπάρχουν απαντήσεις. Πρέπει να δράσουμε για να προλάβουμε την επανάληψη νέων καταστροφών ανθρωπιστικής φύσεως και να αποφύγουμε την, τη σπατάλη μια νέα γενιά ακόμα, η οποία απλώ θέλει ένα καλύτερο αύριο. Η διεθνή κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνουν όλου του φορεί στο διάλογο και στη διεύρυνση του χώρου ελευθερία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη θα πρέπει να συνοδεύσουν και να υποστηρίξουν τι χώρε αυτέ για να διεξάγουν ελεύθερε και αξιόπιτες εκλογές. Το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα μπορούσε να συνεισφέρει στις προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών στο Κονγκό για να εξασφαλίσουμε την παρακολούθηση και την αφύπνιση σε μία άσκηση δημοκρατικού δικαιώματος. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό η διακυβέρνηση είναι προτεραιότητα και οι αρχές της χώρας με την υποστήριξη των διεθνών φορέων θα πρέπει να δεσμευτούν πολύ συγκεκριμένα να βελτιώσουν τη διαφάνεια κατά τη διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων και να καταπολεμήσουν τη διαφθορά. Πριν από δύο εβδομάδες, λαμβάνοντας την έκθεση του Ειδικού Συμβούλου του Προέδρου της Δημοκρατίας που μιλούσε για την ε, διασπάθηση χρήματος, για τη διαφθορά και για το ότι έχασε η χώρα 15 ε, δισεκατομμύρια δολάρια από έστω που θα πρέπει να είχε εισπράξει πέρυσι, τίθονται πάρα πολλά ερωτήματα για το τι μπορούμε να κάνουμε όταν υπάρχει τέτοια διαφθορά, τέτοια διαστάθηση χρήματος, τέτοιες λαθροχειρίες. Η καταπολέμηση της διαφθοράς λοιπόν είναι πυλώνας, ε, μια προϋπόθεση για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε συνθήκες ανάπτυξης χωρίς συγκεκριμένες προσπάθειες για να βελτιώσουμε την κατάσταση της ασφάλειας, την δημοκρατική διακυβέρνηση, την αναπτυξιακή, η αναπτυξιακή βοήθεια δεν θα μπορέσει ποτέ να ενισχύσει τους θεσμούς, ούτε να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής του πληθυσμού και ακόμα λιγότερο να συνεισφέρει στις προσπάθειες πολεμηση της στόχης. Αυτή η αναπτυξιακή βοήθεια απλώς εξυπηρετεί κάποια άτομα και καθόλου το μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Κυρίε και κύριοι ευρωβουλευτέ, στην ομιλία που εκφωνήθηκε στο Στρασβούργο κατά την, όταν δόθηκαν τα βραβεία Σαχάροφ, είχα, κατά την μου αυτή είχα πει ότι ε, θα πρέπει η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό να χρησιμοποιήσει τους πόρους, τόσο ανθρωπιστικούς όσο και υλικούς, για να περάσει στην ανάπτυξη. Η χώρα μου πάντα ήταν ένα, ε, μια προϋπόθεση, ένα στοιχείο και μια χώρα που υποβοήθησε την παγκοσμιοποίηση και την εξέλιξη ε, στη σύγχρονη εποχή. Από το Καουτσούκ που επέτρεψε την βιομηχανική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας, το ουράνιο, το οποίο βοήθησε για να τεθεί τέλος ε, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κασίτερο, το βολφράμιο, το ταντάλιο, ε, που έχουν δημιουργήσει επανάσταση στον τρόπο που επικοινωνούμε. Το Κονγκό πάντα ήταν στο κέντρο της πρόοδου. Αλλά δυστυχώς αυτή η πρόοδος ποτέ δεν ήταν η δική μας πρόεδρος, πρόοδος. Ποτέ δεν τη μοιραστήκαμε. Αυτοί οι πόροι που θα μπορούσαν, που επιτρέπουν την πρόοδο της Ευρώπης και τον υπόλοιπο κόσμο, ποτέ δεν ε, βοήθησαν στην ανάπτυξη της χώρας μου και ποτέ δεν ευνόησαν τον κοκολέζικο πληθυσμό πέρα από κάποιους ηθήνοντες και κάποιους ε, ε, επιχειρηματίες που είναι πραγματικά λαμόγια. Σήμερα μπορείτε να συνεισφέρετε για να γραφτεί μια νέα σελίδα της ιστορίας του Κονγκό που να βασίζεται σε συναλλαγές που θα είναι επικερδής αμοιβαία και μια κατάσταση win-win. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν όχι μόνο μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ένα από τους στόχους που εμπνέουν τις, τις εξωτερικές της σχέσεις, με την προώθηση της ε, ανάπτυξης και της ε, ειρήνης και την ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Με κάθε ταπεινοφροσύνη επαναλαμβάνω σήμερα την έκκλησή μου προς τους ερετούς άρχοντες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ των οικονομικών πολιτικών πολιτικών συγγνώμη, και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να θέσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στο κέντρο των οικονομικών σχεδιασμών και χρηματοπιστωτικών σχεδιασμών. Είναι μια ιστορική ευκαιρία για να σπάσει ο φαύλος κύκλος με το εμπόριο των μεταλλευμάτων αίματος. Ε, αυτή η χρυσή ευκαιρία θα παρουσιαστεί στην επόμενη ολομέλεια του Κοινοβουλίου στο τέλος του μήνα. Πρόκειται για μία από τις βασικές αιτίες των κατ' συγκρούσεων και των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως είναι η σεξουαλική, η βία σε μεγάλη κλίμακα που τα θύματα του τα, τα περιθάλπουμε στο νοσοκομείο του Πάντζη. Η υιοθέτηση τη μια υποχρεωτική νομοθεσία για το εμπόριο των μεταλλευμάτων θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ευθυγραμμιστεί με του κανόνε του ΩΣΑ σε ό,τι αφορά τον εφοδιασμό καθώ και τι ε, ε, υποχρεωτικού κανόνε που υιοθετήθηκαν από τι ΗΠΑ και, και πολλές αφρικανικές χώρες μεταξύ των οποίων και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Επίση θα στείλει ένα σαφέστατο μήνυμα στον κόσμο των επιχειρήσεων ε, ότι υπάρχει διαφάνεια. Μα ανησυχεί το γεγονό όμως ότι ο κανονισμός που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ αδύναμος για να επιτρέψει πραγματική αλλαγή. Γιατί επιτρέπει την ε, επιλογή στους εισαγωγείς να προμηθευτούν αν θέλουν με υπεύθυνο τρόπο ή αν δεν θέλουν με μη υπεύθυνο τρόπο τα μεταλλεύματα αυτά. Ο εθελοντικός μηχανισμός αφορά το 0,05% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν αυτά τα μεταλλεύματα στο Ευρωπαϊκό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, εάν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υιοθετηθεί, καμία επιχείρηση δεν είναι νομικά υποχρεωμένη να επαληθεύει εάν συμμετέχει στη χρηματοδότηση συγκρούσεων ή στην παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα μέτρα λογικής επαγρύπνησης, τα υποχρεωτικά, αφορούν δυστυχώς μόνο τις 20, τα 20 χιτευτήρια και διηληστήρια ε, αυτών των τριών μεταλλευμάτων και του χρυσού στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε όμως νομική δέσμευση που θα αφορά όλες τις ε, επιχειρήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μεταλλεύματα και να μην αφορούν μόνο μία φούχτα από χιτευτήρια. Θα πάμε ακόμα πιο μακριά. Σας καλούμε να στηρίξετε και να ενισχύσετε τους μηχανισμούς πιστοποίησης που έχει θεσπίσει η Διεθνή Διάσκεψη της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών για να γίνεται μία εξόριξη των μεταλλευμάτων που να σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Όταν βλέπουμε παιδιά σε αυτά τα ορυχεία, Ξέρουμε ότι οι γυναίκες φεύγουν από τα σπίτια τους για να πάνε να δουλέψουν εκεί, σε αυτές τις περιοχές. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η πιστοποίηση να γίνεται, ούτω ώστε η εκμετάλλευση να γίνεται με διαφανή τρόπο, να μην μπαίνει στο παιχνίδι ο στρατός. Υπάρχουν περιοχές όπου οι ένοπλες κρατικές δυνάμεις έχουν τον έλεγχο των εκμεταλλεύσεων αυτών. Αν είχαμε όμως μια τέτοια πιστοποίηση, όπως αυτή σας προανέφερα, θα ξέραμε ποιες είναι οι ζώνες όπου γίνεται σωστή εκμετάλλευση και ποιες είναι αυτές που δεν γίνεται σωστή. Ο πρώτος κλίκος αλυσίδας ανιχνευσιμότητας, αν αυτός ο πρώτος κύκλος είναι βρώμικος, το τελικό προϊόν που καταναλώνουμε κάθε μέρα, και αυτό θα είναι στιγματισμένο από το αίμα των γυναικών του Κονγκό. Πρέπει τα λόγια αυτά να τα κάνουμε πράξεις και να κινητοποιήσουμε όλη την ενέργεια και τη θέληση που έχουμε για να φτάσουμε σε μια ειρήνη και μια βιώσιμη ανάπτυξη στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας είμαι πολύ ευγνώμων που ήρθατε να με ακούσετε Δευτέρα απόγευμα. Αγαπητέ γιατρέ, μας δώσατε μια γενική εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Δημοκρατία του Κονγκό και οι χώρες της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών. Είμαι σίγουρη πως οι συνάδελφοι έχουν πολλές ερωτήσεις. Ο κύριος Στίερ, πρώτος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε δόκτορα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ πέρα και το Σάββατο όταν ε, και συζητήσαμε τον ρόλο των γυναικών στην ανάπτυξη αλλά και σας ευχαριστώ για την δουλειά που κάνετε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που πραγματικά είναι ηρωική και την οποία τιμούμε σωστά επισημάνατε το βασικό ζήτημα της ε, ανάπτυξης όταν αναφερθήκατε στην ποιότητα των θεσμών πολιτικών ε, και οικονομικών της ε, χώρας σας και αυτό έχει μεγάλη σημασία και για το ΕΛΚ και για τις άλλες ομάδες του Κοινοβουλίου περάσαμε ένα νέο ψήφισμα το οποίο επισημαίνει ακριβώς αυτό το θέμα το οποίο είναι στον πυρήνα της υπόθεσης γιατί πρέπει να δούμε τα θέματα διαφθοράς παρανόμων χρηματικών ροών και ζητήσαμε και από την Κομισιόν μια ανακοίνωση για τα θέματα αυτά. Επίσης αναφερθήκατε και στα μεταλλεύματα από περιοχές συγκρούσεων όπως ξέρετε το Κοινοβούλιο ε, στις διάφορες επιτροπές του έχει φέρει το θέμα της υποχρεωτικής πιστοποίησης. Βεβαίω τίθεται το θέμα του εύρους, αλλά βλέπετε πως υπάρχουν κάποιες, κάποια κίνηση σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν και μια συζήτηση η οποία συνεχίζεται. Αλλά τελικά θα δούμε και το πώς λειτουργούν οι θεσμοί και πώς συνεισφέρουν στην ορθή διακυβέρνηση, στο κράτος δικαίου, στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, στη συνεργασία με εσάς και με αυτούς που προάγουν τις δημοκρατικές αρχές στη χώρα. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω πως η ομάδα μας υποστηρίζει πλήρως αυτές τις προσπάθειες και να πω πως ακούσαμε όλα σας τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε και πάλι για την δουλειά που έχετε κάνει. Σας ευχαριστώ κύριε Στίερ. κυρία Σίλβα Περέιρα έχει το λόγο για τους ε, σοσιαλιστές. Ο κύριος Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με βάση αυτά που είπε ο προηγούμενος ομιλητής, A intervenção euh, euh, Και έχοντα ακούσει τον δόκτωρα Μουκουέγγε, πρέπει να πω ότι όπως πάντα ήταν εμπνευσμένο και πιστικός ο λόγος του. Μας είπε καταρχήν ναι. ότι όλοι οι δείκτες βρίσκονται στο κόκκινο και πράγματι στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και στην περιοχή των μεγάλων λιμνών είναι πολύ δύσκολο να δει κανείς σε τι να ανταποκριθεί πρώτος. Υπάρχει το δικαίωμα των δικαιωμάτων των γυναικών, το δικαίωμά τους στην υγεία και στη ζωή. Υπάρχει όμως και η προτεραιότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ασφάλεια, η πολιτική κατάσταση, η διαφθορά. Ακούγοντας τον κύριο Μουκουέγγε, είδα ότι μπροστά σε όλα αυτά τα προβλήματα παρόλα αυτά δεν ε, ξεφεύγει από τον κύριο στόχο του και μας ενθαρρύνει να δούμε τα πράγματα δομημένα και στη ρίζα τους. Αυτό είναι κάτι που δεν συνηθίζουν οι γιατροί και οι διευθυντές νοσοκομείων. Είπατε βέβαια ότι πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω από το απλώς να ανταποκρινόμαστε σε επίγουσες περιπτώσεις. Και η Ένωση πρέπει να διασφαλίσει ότι η πολιτική της εδώ, οι πολιτικές της θα έχουν συνέπεια μεταξύ ανάπτυξης εμπορικών σχέσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει βέβαια επίσης ότι και εμείς πρέπει να τα δούμε σφαιρικά, αποτελεσματικά και με συνέπεια. Εξ ονόματος των σοσιαλιστών λοιπόν θα ήθελα να πω ότι ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να έρθει στο ύψος των περιστάσεων και να μπορέσει να εγκρίνει έναν κανονισμό για τις πιστο, το σύστημα πιστοποιήσεων, υποχρεωτικό σύστημα, δεσμευτικό και όχι αυτοπιστοποίηση Πρέπει αυτό λοιπόν να γίνει και μάλιστα αποτελεσματικά έτσι ώστε ο κάθε κρίκος της αλυσίδας της παραγωγής και διάθεσης των μεταλλευμάτων ας πούμε θα γίνονται όλα σωστά. Άρα για μας είναι προφανείς οι προτεραιότητες. να μην βλέπουμε μόνο το γράμμα του νόμου αλλά και κατά πόσον εφαρμόζεται. Εδώ πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει υποχρεωτικό δεσμευτικό σύστημα πιστοποιήσεων που θα αφορά όπως το ξαναείπα όλους τους κρίκους της αλυσίδας της παραγωγής και διάθεσης των μεταλλευμάτων ώστε και από την άλλη να εφαρμόζονται και όλα αυτά. Αυτή είναι για μας η τρομερή πρόκληση. αλλά όχι μόνο για μας και για τις αρχές της χώρας. Πώς βλέπετε λοιπόν το θέμα της εφαρμογής νέων κανόνων με στόχο να διευθετηθεί το σύστημα της εμπορίας των μεταλλευμάτων. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε ο νόμος θα εφαρμόζεται κιόλα. Ευχαριστώ κυρία Σαρδεντίνη για τους πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ δόκτωρα που ξαναήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκτιμώ την καθαρή σας στάση για τα όρικτα από περιοχές ε, πολέμου και θα πω κάτι για τους συναδέλφους η ιδέα τώρα ότι το Κοινοβούλιο θα περάσει δεσμευτική νομοθεσία δεν ισχύει. Επισημάνατε πως η πρόταση που είναι επιτάπητος αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή Εθνούς Εμπορίου περιορίζεται σε 20 ε, διηληστήρια και χιτήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ μηχανήματα όπως αυτό ε, το κινητό μου δεν παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να δούμε κάποιους κανονισμούς ε, και για τα τελικά αγαθά για να μπορούμε να δούμε τι γίνεται επί τόπου. Εγώ είχα την ευκαιρία πριν από δύο χρόνια να πάω στο Βόρειο και τον Νότιο Κίβου. Είδα τις συνθήκες εργασίας, είδα το τίμημα που πληρώνουν οι άνθρωποι για ένα κιλό κασίτερου και το ότι δεν μπορούν να κάνουν το σωστό, δηλαδή να κάνουν εμπόριο μέσω των επισήμων διόδων ε, θα τους απέφερε λιγότερα κέρδη και είστε πραγματικά μια χώρα με τεράστιο πλούτο που θα έπρεπε να ε, εκμεταλλεύεστε. Σας παρακαλώ λοιπόν βοηθήστε μας να βρεθεί ο σωστός τρόπος να σπάσει αυτή η κατάρα πλέον που είναι η φυσική πόρη. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω τις τελευταίες εβδομάδες ε, έχει αποδείξει ότι θέλει να σταματήσει τον πόλεμο στο Ανατολικό Κονγκό. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιο άλλο τον λόγο. Δεν έχουν δώσει άλλο νόμο. Το κύριο Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον δόκτορα Μουγβέγκε για την παρουσία του ακόμα μια φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τη δέσμευσή του απέναντι στις ε, διοκόμενες γυναίκες και απέναντι στους στοχούς της περιοχής αυτής ε, του πλανήτη, των μεγάλων λιμνών και εν γέννη ε, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Μου έκανε εντύπωση η αναφορά που κάνατε για, την, τα θέματα της ασφάλειας στις ε, πολιτοφυλακές ΑΝΤΕΕΦ Ναλού που συνδέονται με το τζιχαντιστικό κίνημα Πιστεύετε ότι η επιρροή τους μπορεί να επεκταθεί σε όλη την περιοχή, πέρα από το Κονγκό. Επίσης, ως στοιχείο της αστάθειας αναφέρατε ότι είναι η επανεκλογή συγκεκριμένων προσώπων στην Προεδρία διαφόρων χωρών. Μέσα σε λίγες μέρες θα πάω στην Μπουζουμπούρα, στις 24 του μηνός, για τις πρώτες εκλογικές αναμετρήσεις που θα γίνουν στο Μπουρούντι. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η αντίδρασή σας σε αυτά τα δύο σχόλια που μόλις έκανα για το θέμα την, της ασφάλειας και για το άλλο θέμα της επανεκλογής των ιδίων ατόμων. Ο κ. Γκέρεντς. Ευχαριστώ. Έχω μία πολιτική ερώτηση να θέσω στον δόκτωρα Μουκβέγγε, τον οποίο ευχαριστώ που ήρθε εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πρόβλημα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ως φορέα ανάπτυξη. Είναι το εξή. Εγώ το βλέπω, όπως το βλέπω από τις Βρυξέλλες βέβαια, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της θα πρέπει να δουλέψουν στα πλαίσια μιας εταιρικής σχέσης. Θα πρέπει να σεβαστούν τον συνομιλητή τους, που είναι η κεντρική αρχή της χώρας με την οποία συνεργάζονται. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποια όρια που πρέπει να τεθούν από τις αρχές του Κονγκό σε δράσεις που θα μπορούσαν να αναπτύξουν οι κράτες μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κονγκό. Και μια δευτερεύουσα ερώτηση. Όταν οι θεσμική φορείς, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη-μέλη, δεν γίνονται δεκτά, δεν τα δέχεστε. Τι θέση έχουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις για να υποκαταστήσουν την ε, δράση των φορέων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν γίνονται δεκτοί. Ο κ. Βέντερ ήταν εισηγητής για μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή Ανάπτυξης για, την, ε, για τα μεταλλεύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. μου να πείτε, δόκτωρα Μουκβέγγι, εγώ παρακολουθώ τις ε, δηλώσεις σας και όπως είπε η Πρόεδρος είμαι εισηγητής εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εδώ προσπαθούμε να βρούμε λύσεις ε, που θα είναι ικανοποιητικές και για εσάς. Γιατί εκπροσωπείτε τη χώρα σας εδώ πέρα. Εδώ μιλάμε συνεχώς για υποχρεωτική και εθελοντική πιστοποίηση. Θεωρείτε πως χρειάζονται περαιτέρω βήματα για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια πολιτική σταθερότητα στο Κονγκό, γιατί αυτό είναι ένα σημαντικός παράγοντας για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο των ορυκτών από πολέμους. Ό,τι μπορέσετε να πείτε θα μας βοηθήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπεθέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε δόκτωρα Μουκβέγγε ξανά. Χαίρομαι που σας ευχαριστώ έτσι πρόσωπο με πρόσωπο για τη δέσμευσή σας, γιατί νομίζω ότι κάντε τη δουλειά για την οποία σας δώσαμε το, και το βραβείο Ζαχάρου και σας ευχαριστώ για αυτό. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της πιστοποίησης των μεταλλευμάτων από ζώνες πολέμου και πρέπει να πάρουμε θέση. Και πρέπει να γίνει υποχρεωτική αυτή η πιστοποίηση. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντική δε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη όλη την αλυσίδα παραγωγής, όλα τα βήματα, για να μπορέσουμε να αναχθούμε ως την προέλευση αυτών των μεταλλευμάτων. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτά τα τελικά βήματα που πρέπει να κάνουμε εν ώψη της διαπραγμάτευσης ε, της συμφωνίας TTIP με τις, Ευρω... με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν μια νομοθεσία οι Ηνωμένες Πολιτείες πολύ πιο απαιτητική αυτό το πλαίσιο διαπραγμάτευσης ε, καλό δεν θα ήταν να εναρμονιστεί και να εξισορροπηθεί ούτω ώστε η ικανότητα δράσης που έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως μείζον δωρητής ε, να υποφεληθεί από αυτή τη διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ και να φτάσουμε τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τις ΗΠΑ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλον να ζητάει το λόγο. Δεν ξέρω, η, η Κομισιόν η Υπηρεσία Εξωτερική δράση έχει κάτι να πει από τη Γενική Διεθνή Εμπορίου κύριο ε, Σινιαράτσο η κυρία Σινιαράτσο δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι εδώ το όνομά σα μου πάσαραν Α, όχι, με συγχωρείτε θα σας αφήσουμε στην ησυχία σας. Εντάξει, δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Θα συζητηθεί το θέμα των ορυκτών στην Ολομέλεια και στις Επιτροπές. Ερωτήσεις ε, για τους αρμόδιους για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν υπήρχαν. Κυρία Τισά, όχι, όχι, δεν υπήρχε κάτι για σας. Αυτά. Λοιπόν, έχω εγώ μια ερώτηση, αγαπητέ γιατρέ. Όταν ήρθα εγώ στο Κονγκό, στο νοσοκομείο σας, ε, να σας πω, το να πάει κανείς εκεί πέρα είναι πραγματικά προνόμιο. Δεν είναι απλά ένα νοσοκομείο το οποίο ασχολείται με γυναίκες και παιδιά που είναι θύματα σεξουαλικής βίας, αλλά είναι μια όαση ειρήνης και ελπίδας στην περιοχή. Και βλέπετε πως ο κόσμος το βλέπει ως ένα μέρος ε, ένα πρότυπο διαφορετικού Κονγκό. Φτάνει κανείς και βλέπει μεγάλες συνακίδες που λένε η λαβεριτέ πείτε την αλήθεια» για να πούν το τι τους ε, συνέβη, για να βρεθεί ένας ε, νέος ε, τρόπος για το μέλλον. Και μετά μιλήσατε για την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά βεβαίως η ανθρωπιστική βοήθεια, όπως ξέρουμε, υφίσταται περικοπές. Προσπαθούμε εδώ να διατηρήσουμε τον προπολογισμό της και εσείς θα θέλατε χρηματοδότηση από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης γιατί η ΕΚΟ έχει μόνο ετήσια χρηματοδότηση και για να προγραμματίσει κανείς μακροπρόθεσμα χρειάζεται την ανάλογη χρηματοδότηση. Και οπωσδήποτε εγώ συναντήθηκα με τον Επιτροπο Νίμητσα και του είπα να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Ε, αν θέλετε να μιλήσετε γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να το κάνετε, αλλά είμαι σίγουρη πως και η Επιτροπή μας μπορεί να το δει, γιατί είμαστε υπεύθυνοι και για την ε, χρηματοδότηση της ανάπτυξης και την ανθρωπιστική. Και οπωσδήποτε δεν μπορούμε να αφήσουμε το νοσοκομείο χωρίς ε, χρηματοδότηση. Λοιπόν, Δόκτωρα, δεχτήκατε πολλές ερωτήσεις, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να απαντήσω σε όλα αυτά θα αρχίσω με το βασικότερο ερώτημα διότι Είπατε ότι δεν μίλησα ως χειρούργος. Μάλιστα, σωστό. Αλλά αυτό που μας οδήγησε να θέσουμε τα ερωτήματα που θέτουμε είναι μια καθημερινή εμπειρία. Όταν αρχίσαμε να φροντίζουμε τα θύματα των σεξουαλικής βίας πριν από 15 χρόνια, ως χειρουργοί το κάναμε. Μέχρι τις 10 το βράδυ δουλεύαμε στα χειρουργεία και είχαμε αποτελέσματα. Όταν όμως η ίδια ασθενής που είχατε χειρουργήσει έρχεται για δεύτερη φορά, τότε τι να πείτε. Αν την πρώτη φορά μπορείτε να τη ρωτήσετε γιατί, τι έγινε, τι χειρουργείτε, διορθώνεται ότι είχε καταστραφεί, αλλά για τη δεύτερη φορά δεν υπάρχει πια τίποτα και το μόνο που μπορούμε τότε να πούμε είναι δεν γίνεται τίποτα. Εκείνε απαντούν όχι δεν θα φύγω από το νοσοκομείο αν δεν με βρείτε λύση. Μέχρι τη μέρα που έρχεται να με δει και το παιδί που προήλθε από το βιασμό. Είχε έρθει η γυναίκα, τη βοηθήσαμε στη Χένα και αυτή τη φορά έρχεται με το μωρό, πάλι βιασμένη τότε κατάλαβα ότι κάτι έπρεπε να γίνει κατεπηγόντως. Αφού λοιπόν τα προβλήματα είναι κατεπήγοντα, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά δεν λύνουμε το θέμα της ουσίας, τη ρίζα του κακού. Τότε άρχισα να εγκαταλείπω το χειρουργείο για να σας μιλώ με σας που παίρνετε τις αποφάσεις για να σας πω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που διαθέτουμε και αλλιώς τα χρήματα της ανάπτυξης αλλιώς όχι μόνο για να αντιμετωπίσουμε κατεπίγουσες κατεπήγοντα περιστατικά γιατί έτσι θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση και τώρα συνδέω με την τελευταία ερώτηση έχουμε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΚΟ για πάνω από 10 χρόνια αλλά αυτό είναι αντιμετώπιση κατεπήγουσων καταστάσεων Σήμερα έχει αρχίσει να μειώνεται η βοήθεια αυτή, αλλά δυστυχώς ο αριθμός των θυμάτων δεν μειώθηκε. Και άρα δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μόνο με τα κατεπήγοντα περιστατικά, να βρούμε και άλλες λύσεις. Σήμερα στο νοσοκομείο, όπως είπε και η πρόεδρος, έχουμε μείωση του προϋπολογισμού. Και το πρόβλημά μας είναι ότι πρέπει να επιλέξουμε ποιον να θεραπεύσουμε πολύ δύσκολο δεοντολογικά. Αν έρθουν δύο πελάτησες, δύο ασθενείς, η μία με ακράτεια ούρων και πρέπει να θέσουμε το ερώτημα πώς έγινε αυτό και μου απαντήσουν έγινε μετά από βιασμό δέχεστε να τη φροντίσετε αν όμως είναι μετά από γένα που δεν έγινε όπως έπρεπε και εγώ τη θεωρώ και αυτήν βία πρέπει να μπορέσει η γυναίκα αυτή να θεραπευτεί σωστά. Μου λένε δεν μπόρεσα να γεννήσω σε κανονικές συνθήκες και γι' αυτό καταστράφηκαν τα γεννητικά μου όργανα. Και τότε είμαι αναγκασμένος να πω ότι δεν μπορώ να την αναλάβω. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για έναν γιατρό. Ενώ έχουν το ίδιο πρόβλημα δύο γυναίκες, αποκλείονται κοινωνικά και στιγματίζονται από την κοινωνία. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε στην ανάπτυξη και τη φροντίδα αυτών των γυναικών χωρίς άνηση μεταχείριση Επίσης όμως και την καταπολέμηση της παθολογίας για να μην επαναληφθεί. Και αν δεν έχουμε αυτή τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μπορέσουμε να τα αναλάβουμε όλα αυτά ισότιμα. Το δεύτερο ερώτημα αφορά πολύ περισσότερο τη ρίζα του κακού και τι εννοώ με αυτό. Διοπιστώσαμε ότι τα κύριά μας προβλήματα είναι, προέρχονται από βία σε περιοχές σειράξεων. Αν λοιπόν δεν βρούμε μια απάντηση για αυτό στις σειράξεις θα συνεχίσουν τα ίδια φαινόμενα. Αυτό μας οδήγησε ας πούμε να ενδιαφερθούμε για τα θέματα της ασφάλειας. Είναι ουσιώδης αυτή η μεταρρύθμιση. Αν δεν γίνει σε βάθος θα συνεχίσουν τα ίδια προβλήματα και φαίνεται και σήμερα. Το κακό που έγινε στις περιοχές σειράξεων όταν συνήθισαν οι ειρηνευτικές συμφωνίες αλλά δεν λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι οι ένοπλες ομάδες έχουν ε, ασκήσει προπαγάνδα στους νέους δεν μπορεί να αναλυφθεί καταλήλως η ψυχολογική τους θεραπεία. Μπορεί να έχουν παρατήσει τα όπλα οι νέοι, αλλά πρέπει να θεραπευτούν και διανοητικά. Αλλιώς θα συνεχίσουν τα προβλήματα. Πρέπει το κακό να το χτυπήσουμε λοιπόν στη ρίζα δηλαδή να γίνει μια μεταρρύθμιση που να λαμβάνει υπόψη της και το παρελθόν όσων μπαίνουν στο στρατό, στην αστυνομία για να μπορέσουν να παίξουν σωστά το ρόλο τους για την προστασία της κοινωνίας των πολιτών. Αναλύοντας λοιπόν τους λόγους βλέπουμε ότι τα ορυκτά δεν είναι ο μόνος λόγος των σειράξεων αλλά επιτρέπουν την διατήρηση των σειράξεων. Γιατί τα πολεμοφόδια κοστίζουν, τα όπλα κοστίζουν. Το να, συντηρούμε, το να συντηρηθούν αυτές οι ένοπλες δυνάμεις θέλει. χρειάζονται λεφτά. Και από πού έρχονται αυτά τα λεφτά, που προέρχονται από αυτά τα μεταλλεύματα. Θεωρούμε ότι αν σήμερα οι Ευρωπαίοι βουλευτές όλοι μαζί, δεν μιλάω για καμία συγκεκριμένη πολιτική ομάδα, είναι θέμα ανθρωπιά. Νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτά τα όρια, πρέπει να ξεπεράσουμε τα όρια των πολιτικών ομάδων και να μιλήσω ε, για το, τα αισθήματα που όλοι μοιραζόμαστε. Την, ε, είναι θέμα ανθρωπιά. Αν όλοι καταλαβαίνανε τη σημασία ε, αυτού, του θέματος της αλυσίδας ανεφοδιασμού ξεκινώντας από την πιστοποίηση. Αν πιστοποιούσαμε αυτά τα ορυχεία, θα ξέραμε ακριβώς Ποιος μπήκε για να εξάγει, να εξορίξει και υπό συνθήκες. Ποιος χρησιμοποιεί. Και εδώ, εδώ μιλάω για παιδιά και γυναίκες που κάνουν αυτή τη δουλειά σαν σκλάβοι. Κάθε μέρα πληρώνουν και αν δεν πληρώσουν δέχονται απειλές. Μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Αυτό μας πάει πίσω 200 χρόνια. Είναι θέμα σκλαβοπάζαρου, όπου Κάποιο ένοπλο, α πούμε ε, με, το όπλο με την κάνει το όπλο στραμμένο πάνω σου σε υποχρεώνει να μπει στο ρηχείο. Εσείς καταβαίνετε στα έγκατα του ορυχείου αυτού, εξορίσετε τα μεταλλεύματα και του θα παραδίνετε. Χάρη λοιπόν σε αυτή την πιστοποίηση λύνουμε αυτό το θέμα και με την βοήθεια της κοινωνία των πολιτών μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε πολλά. Ε, στη Σαμπούντα είχα μια συνεδρίαση με την, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Για την ε, εξόριξη του χρυσού χρησιμοποιούν ε, υδράργυρο. Ε, τον υδράργυρο αυτό τον πετάνε σε ποτάμια που το χρησιμοποιούν οι ντόπιοι πληθυσμοί. Είναι πρακτικές οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη τον άνθρωπο δεν ασχολούνται καθόλου με τα προβλήματα που δημιουργούν στο περιβάλλον κτλ. Είμαι πεπισμένο ότι οι άνθρωποι ε, από το χωριό αυτό θα έχουν ε, νεφρικέ ανεπάρκειες, οι θα πρέπει μετά να κουράρουμε. Ενώ βάζαμε σήμερα κανόνες και αν λέγαμε δεν υπάρχει πιθανότητα να εκμεταλλεύσετε το χρυσό μέσα σε, με τέτοιε συνθήκε. Με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομούσαμε πολλά που θα ξοδέψουμε αργότερα για την υγεία. Αλλά δυστυχώ κανένα δεν πιστοποιεί, κανένα δεν ελέγχει πώ εξορίζονται αυτά τα μεταλλεύματα. Όλο το θέμα είναι από πού προέρχονται αυτά τα μεταλλεύματα. Εάν γίνει στην πηγή αυτή η πιστοποίηση, τότε οι ντόπιοι τεχνίτες μπορούν να κάνουν και τη δουλειά τους με την εξασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, που είναι η ελευθερία να αποφασίσουν για τη δουλειά που θα κάνουν και να μην κάνουν καταναγκαστικά έργα και θα ξέρουμε όλοι οι υπόλοιποι αν είναι καθαρά αυτά τα μέταλλα. Αν ξεκινήσουμε από την βάση, όλη την αλυσίδα την ελέγχουμε. Επίσης, πιστεύω ότι η προσπάθεια και ζήτηση πάντα θα είναι ίδια. Και μάλιστα υπάρχει και κάτι που δεν καταλαβαίνω. Γιατί Είμαστε αντίθετοι στο να είναι διαφανής αυτή η αλυσίδα. Τα μεταλλεύματα φεύγουν από το ίδιο σημείο πάντα. Και θα φτάσουν στο κινητό τηλέφωνο που έχουμε ανάγκη εμείς. Επομένως, η σχέση προσφοράς και ζήτηση δεν θα αλλάξει. Πάντα θα υπάρχει ζήτηση. Αλλά θα, καλό θα είναι τα προμηθευτούμε αυτά τα μέταλλα απορρικτά, ασφαλή, ούτω ώστε να μην ταλανίζεται και η συνείδησή μου. Εγώ πήγα σε κάποια από αυτά τα ορυχεία. Ε, μου ήταν αδύνατο να κοιτάξω δεύτερη φορά τα παιδιά αυτά που δούλευαν εκεί. Αν ελέγχουμε αυτή την αλυσίδα, μπορούμε όλοι μας να παίρνουμε και καθαρά μεταλλεύματα, χωρίς αίμα δηλαδή, ενώ τίποτα δεν θα αλλάξει. Ενώ σήμερα τι κάνουμε, βοηθάμε αυτές τις εγκληματικές ομάδες να κερδίσουν πάρα πολλά. Το βασικό είναι ότι δεν πρέπει να πληγεί η αγορά μας. Πάντα θα έχει τα μεταλλεύματα που χρειάζεται. Εμείς κάνουμε μία μελέτη στο Πάντζι για να δούμε από πού προέρχονταν αυτές οι γυναίκες που ήταν θύματα και κουράραμε στο νοσοκομείο μας και διαπιστώσαμε ότι οι γυναίκες αυτές προερχόταν από αυτές τις περιοχές όπου υπάρχουν πολλά ορχεία. Αυτές οι, οι ομάδες, ας πούμε, πολεμούν μεταξύ τους για να ελέγχουν αυτές τις περιοχές. Αλλά σήμερα δεν είναι μόνο οι πολιτοφυλακές αυτές, αυτές οι ομάδες, ας πούμε, οι ένοπλες. Το Κονγκό είναι τεράστια χώρα και το ερώτημα είναι γιατί το πρόβλημα βρίσκεται στα ανατολικά του Κόγκο Από την εποχή που υπογράψαμε τις ε, ειρηνευτικές συμφωνίες ε, έχουμε σύγκρουση, ένοπλη σύγκρουση, εκεί όπου υπάρχουν αυτά τα ορυχεία. Από το βορρά μέχρι το νότο του Ανατολικού Κογκό. σε ένα κάθετο άξονα. Και αυτά τα μεταλλεύματα δημιουργούν όλο το πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και το θέμα των εκλογών από την άλλη. Το μεγάλο μας μέλημα σήμερα είναι να υπάρχει μια δημοκρατική εναλλαγή στη λαϊκή δημοκρατία του Κόγκο. Μπορούμε να συγκρίνουμε δύο καταστάσεις. Σήμερα βλέπουμε τι ζούμε στο Κόγκο, τη διαφορά που υπάρχει, την ακυβερνησία που υπάρχει. Σε πολλές περιοχές δεν υπάρχει κρατική εξουσία, είναι ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Και υπ' αυτές τις συνθήκες το μέλλον είναι ζωφερό. Χθες με ρωτήσανε τι γίνεται με το θέμα της μετανάστευσης και εγώ απάντησα ότι αυτό εδώ, αυτό εδώ στην Ευρώπη σας απασχολεί. Είμαι σίγουρος όμως ότι αν θα έχουμε ένα τίμιο εμπόριο που θα επιτρέπει ε, στους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις περιοχές να έχουν και αυτή τη δυνατότητα να δουλέψουν, να κερδίσουν τη ζωή τους να, να έχουν ένα καλό βιωτικό επίπεδο, μπορούν να μείνουν στη χώρα τους και δεν θα παίρνουν το ρίσκο, ας πούμε, να περάσει τη Μεσόγειο και να πνιγεί εκεί. Αλλά οι νέοι μας δεν έχουν ελπίδα πια, έχουν χάσει την ελπίδα, η ανεργία. Η ανεργία ε, είναι απίθανη. Δεν έχει νόημα να ρωτάμε πού, πού δουλεύεις, αλλά το αν δούλεψες ποτέ. Τα διπλώματα δεν αξίζουν τίποτα. Η απάντηση λοιπόν το πρόβλημα τη μετανάστευση θα ήταν να δώσουμε τη δυνατότητα στου νέου αυτούς, εάν θέλουν να δουλέψουν στα ορυχεία, να δουλέψουν, αλλά να κερδίσουν και κάτι για τη δουλειά τους. κάναμε και έρευνε σε ορισμένες περιοχές όπου άνθρωποι ζουν, μια ολόκληρη οικογένεια δηλαδή, ζει με 26 δολάρια το μήνα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες τα παιδιά φεύγουν στη Νότιο Αφρική, φεύγουν προ όλες τι κατευθύνσεις. Σήμερα δεν υπάρχει λύση. Εάν δεν διαφανείς καθαρές εκλογές που θα επιτρέψουν πρώτον να εκφραστεί ο πληθυσμό και θα θέλαμε γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας βοηθήσει, να βοηθήσει την κοινωνία των πολιτών. Να πάνε οι οργανώσεις αυτές να μιλήσουν με τους πολίτες να βοηθήσουν τις γυναίκες που κάνουν πολλά για την κοινωνία μας. Αλλά αυτές οι δραστήριες γυναίκες παραμένουν μόνο σε επίπεδο έτσι, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και δεν πάνε παραπέρα. Γιατί πιστεύουν ότι η πολιτική είναι βρώμικη, ότι δεν είναι για αυτές και καταλείπουν την πολιτική. Ενώ κάνουν μια αξιοθαύμαστη δουλειά στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Και εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μας βοηθήσει για να συμμετάσχουν πολύ περισσότερες γυναίκες στην πολιτική. Και αυτό θα άλλαζε τα πράγματα. Γιατί όταν βλέπουμε τι κάνουν οι γυναίκες στις οργανώσεις, είμαστε πεπισμένοι ότι αν τις τονώσουμε και τις σπρώξουμε για να συμμετάσχουν και στο επίπεδο που λαμβάνονται οι αποφάσεις, αυτό θα κάνει όλη τη διαφορά. Γιατί ήδη για την, την καταπολέμηση της διαφθοράς πιστεύω ότι καλό θα ήταν να μας βοηθήσετε για να σπρώξουμε όσο μπορούμε περισσότερες γυναίκες να πάρουν σημαντικές πολιτικές θέσεις για να βοηθήσουμε τη χώρα μας να βγει από αυτό το μαρασμό και να βγούμε από αυτό το σύστημα διαφθοράς που υποσκάπτει οποιαδήποτε δυνατότητα και δυναμικό ανάπτυξης έχουμε. Πιστεύω ότι απάντησα στις ερωτήσεις. Πράγματι νομίζω το κάνατε και μας δώσατε μια αίσθηση των τεράστιων προκλήσεων που αντιμετωπίζετε πριν. Τελειώσουμε. Θα δώσω τον λόγο στον Λουί Μισελ. Έχετε κάποια σχόλια. Έχουμε λίγα λεπτάκια ακόμα. Ναι, αλλά θα είμαι πολύ σύντομο. Φυσικά υποστηρίζω αυτά που είπε ο δόκτωρ. Και αυτά είναι και επίκαιρα. Δεν υπόθηκε μένα, αλλά μεταξύ μας υπάρχει ευρεία συνένεση να είναι υποχρεωτικός έλεγχος των μεταλλευμάτων από περιοχές σειράξεων. Και πιστεύω και εγώ όπως και εκείνο ότι αν θέλουμε να γίνει τέτοιος έλεγχος υποχρεωτικός αυτό δεν θα είχε νόημα παρά μόνο αν ίσχυε για όλη τη διαδρομή του μεταλλεύματος. Γιατί αν δεν γίνει σε όλο το βάθος τότε ορισμένες επιχειρήσεις θα θελήσουν να αποκρύψουν την προέλευση του μεταλλεύματος. Σήμερα λοιπόν είναι δύσκολο και στη δική μου ομάδα να πείσουμε όλους τους βουλευτές για τη σημασία που έχει ένας πλήρης έλεγχος σε όλη τη διαδρομή του μεταλλεύματος μέχρι το τελευταίο μεταποιημένο προϊόν. Αλλιώς οι μεταποιητές δεν θα πιστούν να σεβαστούν τον κανόνα της προέλευσης του μεταλλεύματος. Όσοι επισκέπτονται συχνά την Αφρική και γνωρίζουν τα αφρικανικά, όπως νομίζω και εγώ, ξέρουν ότι το θέμα αυτό είναι ουσιώδες για να αποφευχθεί η χρηματοδότηση εμέσως των σειράξεων με τα γνωστά τους αποτελέσματα. Εκείνος βέβαια είναι θεραπευτής και ξέρει τι λέει. Ευχαριστούμε Λουί Μισελ. Ακούγοντάς σας δόκτωρα Μακουέγγι, εμείς έχουμε μια αρχή της αναπτυξιακής πολιτικής που είναι η συνέπειά της δεν θέλουμε σε μια επιτροπή να μιλάμε για την, σε μια επιτροπή μιλάμε για την ανάπτυξη ενώ σε άλλη δεν την επιτρέπουμε. Την επόμενη εβδομάδα νομίζω θα ψηφίσουμε για τα μεταλλεύματα από περιοχές Ιράξεων και πρέπει να τα πούμε αυτά εκεί. Για το άλλο που είπατε τόσο εύγλωτα όπως μου είχατε πει και στο Κονγκό είναι το θέμα της χρηματοδότησης του νοσοκομείου Πάντζη. Θα το θέσουμε και αυτό. Βλέπω την κυρία Ντέρη από το, από το ΕΛΚ και την συγχρηματοδότηση ΕΚΟ και ΝΤΕΒ θα την συζητήσουμε δεν θέλουμε μία γυναίκα να μπορεί να, φρο... να τύχει θεραπείας επειδή έχει βιαστεί, αλλά άλλη όχι επειδή για άλλους λόγους. Πρέπει να βρούμε μια λύση και γι' αυτό επίσης. Εκτός από πρόεδρος της Επιτροπής μας, είμαι και συμπρόεδρος της Επιτροπής για την επιτήρηση των εκλογών. Άκουσα προσεκτικά αυτά που είπατε για την ανάγκη που έχει να υποστηρίξει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό η Ένωση για την προετοιμασία των εκλογών του χρόνου για να δημιουργηθεί κλίμα διαλόγου ώστε να είναι ειρηνικές οι εκλογές και να μην επιστρέψουμε στην κατάσταση του 90. Είναι και άλλοι εδώ συνάδελφοι που είναι μέλη της αντιπροσωπείας για τις εκλογές. Θα το προσέξουμε λοιπόν και αυτό. Σας ευχαριστώ ακόμη μια φορά για την προσέλευσή σας μας δώσατε πολύ τροφή για σκέψη και μας δείξατε ποιες είναι οι ευθύνες μας γιατί καμιά φορά μπορεί να είμαστε απομακρυσμένοι από τα πραγματικά προβλήματα και να μιλάμε για τεχνικές μόνο λεπτομέρειες αλλά πρέπει πάντα να ξέρουμε αν αυτά που συζητάμε έχουν πραγματικά επίπτωση στη ζωή των ανθρώπων. Σας παρακαλώ λοιπόν όλους να, να ευχαριστήσουμε τον δόκτωρο Μακουέγγι ακόμη μία φορά. και πριν κλείσει η συνεδρίαση σας υπενθυμίζω ότι το βράδυ προβάλλονται έργα από τη μονάδα για το βραβείο Σάχαροφ και ένα από αυτά θα αφορά τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό θα έρθει και ο δόκτωρ Μακουέγκε στις 6.30 στο Παρλαμεντάριουμ ή στο Κοινοβουλευτάριον είναι θέματα παιδείας στο Κονγκό στις 6.30 στο κοινοβουλευτάριο Ευχαριστώ πολύ και τους ήρμηνες.